ότι έχει εγκριθεί η ερμηνεία αυτού του άρθρου. Ευχαριστούμε και θα περάσουμε ε, στην ψηφοφορία. Διαδικαστικό έχετε. Κέρβε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, στις 4 Φεβρουαρίου έστειλα πολύ σημαντική επιστολή ε, στον Πρόεδρο, αλλά δεν με τίμησε με απάντηση. Ε, και με αντίστοιχε συζητήσει ε, με διάφορου συναδέλφου από διάφορε πολιτικέ ομάδε ε, είδαμε ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα και επειδή έχουμε 751 τώρα μάρτυρες, τους μάρτυρες, το ξαναλέω γιατί θα τα στείλουμε και πάλι την επιστολή. Γεια Θέλω απλά να επενθυμίσω ότι δόθηκε χθε το βραβείο της Ειρήνης ε, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να τοποθετηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, γιατί υπάρχουν ελπίδες για την ε, δύναμη και την υγεία. Θα περάσουμε τώρα στην έκθεση για Σλοφιέσκα για το πρωτόκολλο της συμφωνίας με την Ελβετία. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Ε, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Σόγκορ, έκθεση Σόγκορ. Τριμερής Κοινωνικής Σύνοδος Κορυφής για την Ανάπτυξη και για την Απασχόληση. Ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση μπέλετε τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοείας. Εγκρίνεται η σύσταση να με τη συμφωνία σε ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Λάμστορφ, ε, έκθεση για τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ε, ε, ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Ονομαστική ψηφοφορία, Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης για την εργασία στον τομέα της αλίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ σε όλους και όλες που συνεργάστηκαν για αυτό το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει θέση υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα πρέπει ε, να ε, ενισχύσει τη θέση των αλλιέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας ε, τα δικαιώματά τους, ψηλότερους μισθούς, κοινωνική στήριξη κλπ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας θα πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να μην θύρονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ε, είναι σημαντικό που εξασφαλίστηκε μια ευρία πλειοψηφία για τα κοινωνικά δικαιώματα των αλλιέων ε, και ελπίζω ότι θα ψηφίσετε θετικά. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην έκθεση για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία. Πρόταση ψηφίσματος από το UNF. E Πρώτα απ' όλα με ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος πέντε πολιτικών ομάδων για το άρθρο 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 4, το πρωτότυπο κείμενο, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, παράγραφος 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 7 ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίστε Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 8. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά το άρθρο 8, η τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ονομαστική ψηφοφορία. Έρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική αναφορά 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται λογική αναφορά 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τη λογική σκέψη α σε δύο τμήματα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λογική σκέψη C σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας G. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας W η πρώτη τροπολογία με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Κατόπιν πρώτο το υποκείμενο ε, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Εκτιμώντας Z, ε, ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές. Πρέπει να γίνει επαλήθευση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. το σύνολο του ψηφίσματος. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Περάς. Κρίθηκε. Θα περάσουμε στην έκθεση Καστάλτο τώρα για τις ε, σχέσεις με την Τουρκία. Παρακαλώ, κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έγινε. Ε, για αυτή την έκθεση, η οποία στοχεύει στο να ενισχύσει τις ε, εταιρικέ σχέσεις, ε, κυρίως με τους σημαντικούς εταίρους που είναι στη Μεσόγειο. Επίση, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερμά τους Τινήσιους και τις τεράστιες προσπάθειες που έχει κάνει η κοινωνία των πολιτών στην Τινησία τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά τους αξίζει το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη και εμείς πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη και κάποια οξυδέρκεια για το μέλλον. Άρθρο 27. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 31. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 34 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 43 υπέρ ε, πρώτο τμήμα συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 50. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία έναρξης ψηφοφορίας. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρθρο 61. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 62. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 64 ονομαστική ψηφοφορία έναρξη λήξη εγκρίνεται Αιτιολογική σκέψη M. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Καστάλ. Έκθεση μπάλα Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 1. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 2. Σε δύο τμήματα. Με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 7. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 8. Σε δύο τμήματα. Με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 11. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ας ε, επιβεβαιώσουμε ονομαστική ψηφοφορία έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Άρθρο 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 15. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 18. Σε έξι τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Έκτο τμήμα έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 22 σε τρία τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 24. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά εποχές. εγκρίνεται. Άρθρο 25. Σε δύο τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 28 σε δύο τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 29. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Έναρξη. Όχι. Επιβεβαιώνουμε έτσι. Επιβεβαιώνουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Άρθρο 30. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Ας επιβεβαιώσουμε και εδώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Άρθρο 31. Σε τέσσερα τμήματα ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 32. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. Άρθρο 35. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 48. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επιβεβαιώνουμε. Ένα εξωφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για επιβεβαίωση. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Άρθρο 49. Νο, ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Άρθρο 51. Ονομαστική ουσιοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 52. Σε πέντε τμήματα όλα με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 53. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Άρθρο 54. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 56. Σε δύο τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 57. Νοονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επιβεβαιώνουμε. Με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Άρθρο 59. Λήξη. Εγκρίνεται. Ε, πρώτη τελική σκέψη. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη D. Τρία τμήματα. Ε, συγγνώμη. Λάθος, κάνω, κάνω λάθος λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, Αιτιολική σκέψη D. Δύο τμήματα. Με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. 16. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ε, Τελική π. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη α, κεφάλαιο α μικρό, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α κεφαλαίο διπεζό, πεζό. Δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σχέδιο ψηφίσματο συνολικά στο σύνολό του ε, η ψηφοφορία. Λυγή. εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπάλας. Ε, για διαδικαστικό θέμα ποιος έχει ζητήσει το λόγο? Ο κύριος Τσανέτσκι. Κυρίες και κύριοι, αν έχει την καλοσύνη με μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά την ε, ψηφορία θέλω να πω το εξής ε, Σήμερα το πρωί υπήρξε ένα επεισόδιο, όχι ε, στο θεωρείο για τους διπλωμάτες. Είχαμε το Ρώσο πρέσβη, τον κύριο Ξούζοφ, στην αίθουσα. Εδώ όμως, ε, λυπάμαι, εδώ δεν είναι η Δούμα της Ρωσίας. Δεν μπορεί ο πρέσβης να μπαίνει εδώ σε μια τέτοια συζήτηση. Και θέλω να επισημάνω κάτι τέτοιο παρακαλώ πολύ να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Εγώ προσωπικά ε, πρέπει να σας πω ότι ήμουν συγκεντρωμένη στην ψηφορία και δεν είδα τίποτα, δεν μπορούσα να δω, αλλά εν πάση περιπτώσει καταγράφουμε αυτό που είπατε. Και κάτι άλλο. Λοιπόν, άλλα δύο διαδικαστικά. Ε, ο συνάδελφός μας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε, εγώ θέλω να μιλήσω για την ψηφοφορία για την έκθεση μόλις ψηφίσαμε μου εισηγητής. Ευχαριστώ τους όδη. Ήταν επαχθή και μακρά η εργασία, αλλά ήταν εξαιρετική. Η Ευρώπη θέλει κοινωνική πρόοδο. Ακούγεται η φωνή του Κοινοβουλίου. Αμέσω αμέργων. Ας το εφαρμόσουμε. Λάμστορφ. Θα ήθελα να τοποθετηθώ πολύ σύντομα σε αυτά που είπε ο συνάδελφος κ. Ζανέτσκι. Έχουμε εδώ κανόνες. Οι διπλωμάτες άλλων κρατών ε, ε, μπορούν ε, να συμμετέχουν στις εργασίες μας σε δύο διπλωμάτες αναπρεσβεία. Είμαστε ανοιχτοί εδώ, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά έκανε ο Ρώσος πρέσβης και ήρθε εδώ και άκουσε τι συζητάμε. Την Κυριακή έχουμε εκλογές στη Δούμα και θα ήταν πάρα πολύ καλό η Δούμα να γίνει εξίσου ζωντανή όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην τελευταία ψηφοφορία. Ε, Κατεξουδότηση κανονισμό τη Επιτροπή για τη συμπλήρωση του κανονισμού 1286-2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα κλπ. Άρθρο 4. Κυρία Περέ. Ευχαριστώ. Κατά πάσα πιθανότητα ε, θα απορρίψουμε την πρόταση για τις τεχνικές προδιαγραφές που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν εισακούστηκαν ε, τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Παραβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την προστασία των ε, λιανοεπενδυτών και για το επίπεδο 2 ε, το περιεχόμενο και γι' αυτό υποβάλαμε αυτή τροπολογία 2. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπερές. Ε, θέλει κάποιο να τοποθετηθεί για αυτή την τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το ψήφισμα, το σύνολο του ψηφίσματος. Χρειαζόμαστε 376 ε, ψήφους ε, για να είμαστε σίγουροι ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχιτε.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 Colleagues, we the to the and I would like... Συνάδελφοι, ε, επεξηγήσεις ψήφου, οπότε όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το κάνουν και να παραμείνουν όσοι θέλουν να κάνουν επεξηγήσεις. Începem Ας αρχίσουμε με τις ε, επεξηγήσεις ψήφου, παρακαλώ. Έχουμε πρώτα απ' όλα την